δούμε σήμερα θα απαντηθούν γραπτώ. Σα ευχαριστούμε, Υπουργέ. Δύο ενημερωτικά στοιχεία. Η συνάντηση στι 5 στις 5 Οκτωβρίου των νομικών υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων αποφάσισε ότι είναι απαράδεκτο η κοινοβουλευτική ασυλία του κυρίου Φιόρε να έρθει. Απόφαση του Ενδένστητο της Ιταλίας ε, από το 2009 στις 24 Αυγούστου από εισαγγελέα της Ιταλίας. Αυτή την απόφαση λοιπόν την μεταβίβασα στην αρμόδια Ιταλική Αρχή. Επίσης από το ομάδες του ΕΛΚ και του ΙΕΦΤΗ έλαβα πολλές ε, αιτήσει για αλλαγέ